για ε, αυτή την εξέλιξη. Την... Σε ευχαριστούμε που είμαστε σήμερα. Ναι, πράγματι. Έχετε δίκιο. Και θα το σημειώσουμε και στα πρακτικά για τη Βασίλη Σελισάβετ. Λοιπόν, να εγκρίνουμε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Υπάρχουν κείμενα, έχετε λάβει όλα αυτά τα κείμενα, υπάρχουν αντιρρήσεις. Αν δεν υπάρχουν, περνάμε σε μια ανακοίνωση.